δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία. Και δίνω αμέσως το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου στον Υπουργό κύριο Βενιζέλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρότι η περιοδική προεδρία του συμβουλίου δεν μετέχει στις συναντήσεις κορυφής που πραγματοποιεί η ευρωπαϊκή ένωση με τη ρωσία ή άλλα τρίτα κράτη έχουμε ε, με χαρά αναλάβει το καθήκον να σας ενημερώσουμε για το τι συνέβη στη σύνοδο κορυφής ευρωπαϊκής ένωσης ρωσίας την προηγούμενη εβδομάδα. η σύνοδος αυτή έδωσε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία προφανώς λόγω της ουκρανικής κρίσης την ευκαιρία να συζητηθούν ανοιχτά θεμελιώδη ζητήματα των σχέσεων της ευρώπης με τη ρωσία. είναι αναγκαίο να μεταδώσουμε το ισχυρό μήνυμα ότι οι πρόσφατες κρίσιμες εξελίξεις πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να τεθεί η εταιρική σχέση μας σε ορθή τροχιά. αυτό αφορά στην ε, διαφορετική προσέγγιση μας ως προς την ανατολική εταιρική σχέση και την ουκρανία αλλά και σε ορισμένα εμπορικής φύσης ζητήματα που αποτελούν σημεία τριβής σημεία που θα μπορούσαν εύκολα να επιληθούν. οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στο πλαίσιο του παγκοσμίου οργανισμού εμπορίου αλλά και αυτές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να γίνονται σεβαστές. από την άποψη αυτή ήταν πολύ χρήσιμος και ο διάλογος που είχαμε στο συμβούλιο υπουργών με τον κύριο Λαυρόφ, αλλά και ο διάλογος που είχαμε στην τελευταία σύνοδο του συμβουλίου εξωτερικών υποθέσεων μόνοι μας οι υπουργοί των κρατών μελών γύρω από τις σχέσεις μας με τη ρωσία. στη σύνοδο πραγματοποιήθηκε ένας ειλικρινής και ανοιχτός διάλογος για αυτά τα θέματα. χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την ετοιμότητα της ρωσικής ομοσπονδίας να μετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση. πιστεύουμε ότι η ρωσία αντιλαμβάνεται τόσο τις προκλήσεις που οι εξελίξεις αυτές ενέχουν για τις σχέσεις μας όσο και το ότι η ίδια έχει ένα ισχυρό συμφέρον να διατηρήσει αυτή τη συνεργασία με την ευρωπαϊκή ένωση σε όσο γίνεται πιο επικοδομητικό πλαίσιο. γνωρίζω ότι ο επίτροπος ο κ. Φίλε, ο οποίος έχει καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες για την ανατολική εταιρική σχέση θα έχει περισσότερα να πει για αυτά τα θέματα και για τα αποτελέσματα των συνομιλιών. επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι και για τις δύο πλευρές είναι σαφής ο βαθμός αλληλεξάρτησής τους η ευρωπαϊκή ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο με απόσταση εμπορικό εταίρο της ρωσίας καλύπτοντας το 45 του συνολικού ρωσικού εξαγωγικού εμπορίου και η ρωσία είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ευρωπαϊκής ένωσης μετά τις ηνωμένες πολιτείες και την κίνα. η ασφάλεια στην κοινή μας ήπειρο και ευρύτερα μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η ρωσία και η ευρωπαϊκή ένωση συνεργαστούν στενά λαμβάνοντας αυτό υπόψη είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκής ένωσης και ρωσίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αξιολογήθηκε θετικά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής και οι δύο πλευρές εκτίμησαν την καλή συνεργασία του στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του ιράν και η ρωσία συνεχάρει την κυρία άστον για την προσωπική της συμβολή στην επιτυχή έκβαση των συνομιλιών ε συν προκειμένου δε να επιτευχθεί μια μόνιμη λύση με το ιράν παραμένει πάντοτε ζωτική σημασίας η συνέχιση αυτής της πολύ καλής συνεργασίας ευρωπαϊκής ένωσης και ρωσίας. όσον αφορά στη συρία συνεργαζόμαστε πλέον πολύ καλύτερα με τη ρωσία ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διάσκεψης γενέβη 2. η ευρωπαϊκή ένωση έδωσε έμφαση στην ανάγκη της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους σύριους πολίτες και αυτό ήταν ένα βασικό σημείο των παρεμβάσεών μας στο μοντρέ των παρεμβάσεων που έκανε και η κυρία άστον και όλοι οι υπουργοί εξωτερικών κρατών μελών που έτυχε να κληθούμε και να μετάσχουμε με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα του οηε στη συνάντηση αυτή. προφανώς η κατάσταση στην ουκρανία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη σύνοδο κορυφής αλλά δεν ήταν το μόνο θέμα. η ρωσία πρότεινε και πάλι τριμερείς συνομιλίες για την ουκρανία αλλά η ευρωπαϊκή ένωση δεν δέχτηκε αυτή την πρόταση γιατί οι διμερείς σχέσεις είναι διμερείς. αποτελεί σημαντική εξέλιξη συμφωνία για την έναρξη διμερών διαβουλεύσεων εμπειρογνωμόνων για την ανατολική εταιρική σχέση και τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου καθώς και για τις πιθανές συνέπειες που έχουν αυτές οι συμφωνίες για τη ρωσική οικονομία. ελπίζουμε πως αυτές οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθεί επικοδομητικός διάλογος μεταξύ ευρωπαϊκής ένωσης και ρωσίας κατά το προσεχές διάστημα ένα διάλογο που θα βελτιώσει τη συνεργασία και την κατανόηση εν ώψη και τη επόμενη συνόδου κορυφή στι 3 ιουνίου στο σότσι. άλλη μια σημαντική εξέλιξη είναι η υιοθέτηση μια κοινή δήλωση για τη συνεργασία στον τομέα τη αντιμετώπιση τη τρομοκρατία. σε αυτήν επαναλάβαμε και οι δύο πλευρέ τη δέσμευσή μα να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση τη τρομοκρατική απειλή βασισμένη στο σεβασμό του κράτου δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. κυρίε και κύριοι βουλευτέ με δεδομένα τα πρόσφατα γεγονότα η σύνοδος κορυφής δεν αναμενόταν να είναι ιδιαίτερα εύκολη ωστόσο είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ως ευρωπαϊκή ένωση με ειλικρίνεια και θεωρώ πως αυτή η ειλικρίνεια υπήρξε και από την άλλη πλευρά. κάναμε συνεπώς μια καλή αρχή για να επαναφέρουμε τη σχέση μας στην ορθή τροχιά. υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνο μέσω της στενής συνεργασίας. έτσι τόσο η ευρωπαϊκή ένωση όσο και η ρωσία έχουμε ένα ισχυρό κοινό συμφέρον να εργαστούμε μαζί. αυτό ασφαλώς και δεν μας αποτρέπει από το να εκφραζόμαστε ανοιχτά όταν αυτό απαιτείται. θεωρώ ότι καταφέραμε να πετύχουμε και τα δύο αυτά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας. σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. λόγο Uh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω το σώμα για την δεύτερη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ρωσίας που έγινε τον Ιανουάριο στη Ρωσία, στην ε, Βρυξέλλες, με συγχωρείτε. Ήταν μια σημαντική στιγμή. Ο πρόεδρος ο Ρομπόη και ο πρόεδρος Μπαρόζο κατέστησαν σαφές ότι δεν μπορούσε να είναι μια συνηθισμένη συνεδρίαση. Αντί αυτού θέλησαν να εστιάσουν σε μια ειλικρινή συζήτηση για το νόημα και την κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής εταιρική σχέσης. Η διάσκεψη κορυφής περιλάμβανε μια περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη, ένα γεύμα με την είπατε εκπρόσωπο Άστον και τον Υπουργό Εξωτερικών Λαυρόφ, καθώ και μια συνέντευξη τύπου. Τρία θέματα κατέστησε σαφή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη αυτή τη ειλικρινού ε, διάσκεψη. Πρώτον, η ρωσική πίεση στου ανατολικού μα εταίρου είναι απαράδεκτη. Οι κοινοί μα γείτονε θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν οι ίδιοι για την πολιτική και οικονομική Ένωση που θέλουν να συνάψουν, η συμφωνία που θέλουν να συνάψουν. Η Ένωση κατέστησε σαφές πως αναμένει η Ρωσία να σεβαστεί την επιλογή των εταίρων μας και να μην παρεμβαίνει στην υπογραφή των συμφωνιών σύνδεσης ή FTAs με τη Γεωργία ή την Δημοκρατία της Μολδαβίας φέτος. Δεύτερον, μετά από την πρόσβαση της Ρωσίας στον ΠΟΕΔ τον Αύγουστο του 2012 η Ρωσία δεν έχει ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Ανησυχούμε για τον αυξανόμενο αριθμό προστατευτικών εμπορικών μέτρων που πλητούν τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η Ρωσία είναι τώρα παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα. Μαζί με την Τελωνιακή Ένωση, η Ρωσία είναι υπεύθυνη για το 1 τρίτο όλων των προστατευτικών μέτρων που ελήφθησαν το 2013 και για το 1 πέμπτο όλων αυτών των μέτρων που αυτή τη στιγμή είναι ενισχύ. Τρίτον, Υπάρχουν εξαιρετικά πολλές δεσμεύσεις που δεν, ε, πλήρει, ή δεν υλοποιεί η Ρωσία συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να γίνουν σεβαστά, να δημιουργηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ώστε να αναπτυχθεί και να ανθίσει η ε, συνεργασία μας επί τη βάση της στήριξης των δεσμεύσεών μας. Η Ρωσία ήταν έτοιμη να μπει σε μια ειλικρινή και επικοδομητική συζήτηση για αυτά τα θέματα. Επίσης ανέφερε τις ανησυχίες της αλλά και τα ενδιαφέροντα της, ιδιαίτερα γιατί την ενέργεια. Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε πω η Ρωσία δεν είχε κανένα πρόβλημα αρχή με την ανατολική εταιρική σχέση, αλλά ανέφερε διάφορες οικονομικές του ανησυχίες που πραγματικά είναι αμφισβητήσιμες. Συμφωνήθηκε να γίνουν διμερείς διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστούν διάφορα ζητήματα που έθεσε η ρωσική πλευρά σε σχέση με το τι θεωρούν ως δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις των ε, συμφωνιών σύνδεσης ή TFTAs η τη ρωσική οικονομία. Επίσης, συμφωνήθηκε να συνεχιστούν άτυπες διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις για τις δυνατότητες νέας συμφωνίας ανάμεσα στην Ένωση και τη Ρωσία και ελπίζουμε πως θα είμαστε σε θέση να, να, να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις τον το επόμενο καλοκαίρι, τον Ιούνιο, αν υπάρξει αρκετή ουσία για να υπάρξει και νέα συμφωνία. Η Ουκρανία και το Ιράν συζητήθηκαν επίσης και υιοθετήθηκε ένα κοινό, μια κοινή δήλωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστώ. Και πρώτα θα ακούσουμε του ομιλητέ εξ ονόματος των ομάδων. Ο κύριο Μπροκ για ένα μισή λεπτό. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω κάτι ευθύ εξ αρχή. Όσο τα κράτη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μιλούν με μία φωνή στο θέμα της πολιτικής για τη Ρωσία, δηλαδή όσο δεν υπάρχει μία πραγματικά κοινή ρωσική πολιτική θα χάνουμε σε αυτό τον ε, αγώνα. Και αυτό σε συνάρτηση και με την Ουκρανία και με άλλα θέματα και θεωρώ ότι αυτός ε, ο συναγωνισμός αυτό το γεγονός ότι Κάποιοι θέλουν να προηγηθούν και να πηγαίνουν προς τη Μόσχα σε ό,τι αφορά θέματα ενεργειακά και πρωτοσημισιακά δεν ωφελεί κανέναν. Γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα στην τελική ανάλυση και η Ρωσία έχει κοινά συμφέροντα. Ε, αν η Ρωσία έχει μια καλή οικονομική ανάπτυξη και δεν εξαρτάται από την ε, πώληση τέτοιων ε, ε, πρωτονυλών, έχει η Ρωσία, θεωρώ, ευκαιρίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο κοινό συμφέρον το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουμε και από στρατηγικής άποψης. Αυτό τι σημαίνει όμως ότι τη Ρωσία ε, αν θέλουμε ένα νέο τέτοιο στρατηγικό ε, ε πλαίσιο ε, εταιρικής σχέσης θα πρέπει να είναι σαφές ότι τα κράτη τα οποία είναι ανεξάρτητα, είναι ανεξάρτητα αυτό το near broad δεν ισχύει πλέον και δεν επηρεάζονται ούτε από τις Βρυξέλλες, ούτε από το Προλίνο ούτε από τη Μόσχα. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό ισχύει για την Ουκρανία, με την Μολδαβία, η Περνιστερία, Αρμενία. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ενταχθούν σε μια καλή πολιτική γειτονία και η Ρωσία θα πρέπει να αναγνωρίζει επικυρίαρχα κράτη και να τηρεί τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιτρέψει πολιτική αντιπολίτευση. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία. Απέχουμε παρασάγκας όμως από αυτό. Ελπίζω το Σότσι να μην είναι μόνο μία ανάσα, αλλά και ένας τρόπος συνεργασίας σωστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. Εξ στο των ο κύριο Ρούτσεκ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε Υπουργέ. Ακούσαμε ότι έχουμε κοινά συμφέροντα με τη Ρωσία. Είμαστε γείτονε. Η Ρωσία είναι στο Συμβούλιο Ασφαλεία και η κατάσταση στην Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράν με τα πυρηνικά θέματα Όλα αυτά τι καταδεικνύουν ότι υπάρχει ανάγκη συνεργασίας. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώκουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Επιδιώκουμε ένα όραμα κοινής, κοινού οικονομικού χώρου. Αλλά όπως αναφέρθηκε ήδη, επί χρόνια προσπαθούμε να μπει η Ρωσία στον ΠΟΕ. Τώρα, μετά από ένα χρόνο συμμετοχής, βλέπουμε ότι η Ρωσία δεν ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων και στις δεσμεύσεις της, κοιτώντας ε, και τι γίνεται στην ε, γειτονία, ε, βλέπουμε απαράδεκτες πιέσεις να ασκούνται στους γείτονες και βλέπουμε λοιπόν ότι τα θέσαμε αυτά τα θέματα αυτά στη Σύνοδο. Ναι, θέλουμε συνεργασία με τη Ρωσία, θέλουμε να είμαστε στρατηγικοί εταίροι, θέλουμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και να πετύχουμε μια συνεκτική και φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Αλλά αυτό βάσει αμοιβές εμπιστοσύνης. Καταρχάς η Ρωσία θα πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις, να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις από τις συμφωνίες τις οποίες έχει ε, υπογράψει. Και τότε μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ναι, δεν είναι απλή η κατάσταση. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και αμετακίνητα. Εκ παραλλήλου όμως να μην χάσουμε και το όραμα, το στόχο, τον απότερο που έχουμε ε, μπροστά μας, την στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του Άλτε, της Άλντε, ο κύριος Όγιουλάντο, η κυρία Όγιουλάντο, με συγχωρείτε, για ένα μισό λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, θα είμαι πολύ σύντομη. Θα πω μόνο με δύο λόγια ότι οι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία δεν φαίνονται και πολύ καλέ. Ωστόσο, οι σχέσεις μας με τη Ρωσία έχουν χάσει τη δυναμική τους πορεία. Αντί για στενότερους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς, έχουμε διαπιστώσει ότι γίνεται το αντίθετο. Η συνεχιζόμενη επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι απαράδεκτες και μη δημοκρατικές πιέσεις των ανατολικών μας εταίρους, καθώς και η σκληρή ε, παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ, δείχνουν ε, ότι η Ρωσία ε, συνεπώς και συστηματικώς ε, προσπαθεί, ε, μάλλον αναχαιτίζει τη βελτίωση της κατάστασης. Γι' αυτό κιόλας μετεβλήθη η μορφή της διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και η συνεδρία έγινε μόνο για κάποιες ώρες και κλεισμένων των θεωρών αντί να είναι μια διήμερη διάσκεψη κορυφής. Ελπίζουμε ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο και οι εκπροσωποί θα έμεναν στην ίδια συνεπίγραμμα δεν θα πρέπει να ξεγελαστούμε και να πιστέψουμε πως ε, η ξαφνική ε, αυτή ε, παρουσία του Προέδρου θα αλλάξει ή θα βελτιώσει την κατάσταση στη Ρωσία λίγο πριν το Σότσι, ότι θα συνεχιστεί αυτή η στάση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πραγματιστές και να ακούσουμε το λαό της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας που φοβούνται πάρα πολύ οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μετά τους Ολυμπιακούς σε αυτές τις περιοχές Πρέπει λοιπόν όσο γίνεται πιο σύντομα να υπογράψουμε τη συμφωνία σύνδεση με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και προσεχώς και με την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ. Για τους πράσινους ο κύριος Σόλτς για ένα λεπτό. Κύριε Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, δεδομένη και τη συντομία και της, ε, του έντονου χαρακτήρα τη Συνόδου Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία, ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ψήφισμά μα και περιλαμβάνει πάρα πολλά σημεία τα οποία τα έχουμε αναπτύξει εκτενώς και σε άλλα σημεία. Αυτό ίσω να είναι ένα παράδειγμα για το πώ ε, ε, εδώ και πολύ καιρό κινούμαστε μένα, αλλά μένουμε στο ίδιο σημείο. Ίσως να, χρειαζόμαστε, να μην χρειαζόμαστε δύο συνόδου Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία κάθε χρόνο, αν τόσα λίγα έχουμε να πούμε. Ίσως να φτάνει και μία. Θα χρειαζόμαστε μία στρατηγική εταιρική σχέση, δεν την έχουμε όμως. Και το μόνο φετικό της συνόδου αυτή είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν πρότεινε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρική σχέσης. Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει μια ζώνη ελευθερου εμπορίου από τη Λισαβόνα μέχρι το Βαλτιβοστόκ και το ερώτημα το καυτό θα ήταν γιατί μπλοκάρει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου από τη Λισαβόνα μέχρι το Κίεβο. E Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μιγκάλης και από την ΕΣΥΑΡ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Όντω, τρεις ώρες αντί για δύο μέρε πήρε η Σύνοδος Και αυτό καταδεικνύει την ε, κατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας και επίσης καταδεικνύει πόσο άσχημα έχουν πάει τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι το κακό σκέλος, οι κακές ειδήσει. Γιατί είχαμε διαρκή προβλήματα, θέματα ε, όπως στη Συρία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα που μας βρήκαν αντίθετους. Το ψήφισμα που συζητάμε σήμερα δεν τα λαμβάνει υπόψη αυτά επαρκώς. Χαίρομαι που υπάρχουν διάφορα στοιχεία που αναφέρονται, όπως για παράδειγμα η καταδίκη της μεταχείρισης της ρωσικής ζώνης επιρροής σε ό,τι αφορά την μεταχείριση της, ε, ε, των γειτονικών χωρών προς Ανατολά της Ρωσίας. Είναι λοιπόν καλό αυτό που αναφέρετε. Αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, και το άνοιγμα των αρχείων ε, για τις χώρες που άνοικαν στην Σοβιετική Ένωση. Είναι σημαντικό για τα έθνη αυτά. Επίσης, η έκκληση για να μην χρησιμοποιείται η ενέργεια ως πολιτικό ε, όπλο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ξέρουμε ότι η Ρωσία έχει την τάση αυτή να χρησιμοποιεί αυτό το τμήμα της οικονομίας της για πολιτικούς ε, σκοπιμότητες. Και επίσης κάτι άλλο ενδιαφέρον στο ψήφισμα αυτό. Η αντίθεσή μας για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Αυτό όμως που λείπει είναι αυτό που αρχικά αναφέρθηκε από τον Επίτροπο. Θεωρώ ότι είναι πρόβλημα το γεγονός ε, σε ό,τι αφορά τον διορισμό των ομάδων εργασίας που θα εποπτεύουν τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας. Πρόκειται για ένα τέτοιο επιπρόσθετο μέσο το οποίο δεν το καταλαβαίνω με τι νόημα έχει. Βλέπω ότι γνέφεται καταφατικά, Επίτροπε. Απαντήστε μου αν θέλετε. Επίσης δεν αναφέρθηκε τίποτα για το Σότσι. Και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό το πολιτικό μποϊκοτάζ που καθιστά τον Πούτιν ε, δεν επιτρέπει στον Πούτιν να προωθήσει τα συμφέροντά του στο αθλητικό αυτό γεγονός. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος από την ΚΟΕ. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επιτροπέ, ο πρόεδρος του της Επιτροπής Μπαρόσο στη Σύνοδο κάλεσε σε αμοιβή εμπιστοσύνη με τα λόγια του Ντοστοβιέσκη. Καλό ήταν αυτό, αλλά θα έπρεπε να ομολογήσει και στον εαυτό του ότι η λογική της πολιτικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας επί του παρόντος είναι μάλλον η λογική οδόντα αντιοδόντος και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο τώρα και στον τύπο. Η πρόσφατη αυτή σύνοδος ήταν τι να πω, σαν μια ανταπόκριση μεταξύ δύο πτήσεων. Ε, μιλήσανε οι δύο πλευρές, αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι αυτά που δεν συζητήθηκαν. Δεν ε, αναφέρθηκε τίποτα για τα πραγματικά ανοιχτά εκκρεμή ζητήματα, για το φαύλο κύκλο ε, και τις απειλές ασπιδών, Προστασία και πυράβλων. Ήταν λοιπόν αυτή η σύνοδος μια τελέσφορη ε, σύνοδος και αυτό χαρακτηρίστηκε και από σχόλια του BBC. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν ιδέες ό,τι αφορά τους ε, υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαβαίνουμε, όπως λέει ο κύριος Μπρόκ, ότι υπάρχουν αμοιβαία συμφέροντα. Για να μείνουμε στο πλαίσιο του, στο γεύση πρόεδρε, στους αδερφούς Καραμάζοφ τη γράφει ότι ένας ρεαλιστής δεν πιστεύει σε θαύματα όσο δεν είναι πιστός. Τα θαύματα πρέπει να τα δημιουργήσουμε εμείς. Καλό λοιπόν το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το επόμενο, με την επόμενη σύνοδο να έχουν συμφωνήσει σε ένα συγκεκριμένο δικό χάρτη με συγκεκριμένους στόχους. Έχουμε τώρα τον κύριο Στάντλερ. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η σύνοδος αυτή κατέδειξε ένα πράγμα ξεκάθαρα, το οποίο έχει και, ε, προκύψει και τους τελευταίους μήνες. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της ε, Ρωσίας έχει αποτύχει παταγωδός. Και το θέμα της Ουκρανίας. Η Αρμενία κάναμε δεσμεύσεις, υποσχέσεις, τίποτα το συγκεκριμένο και η Ρωσία το ίδιο δεν έχει συμβεί τίποτα τελικά. Είχαμε εδώ πέρα και ένα μέλος της, του Αρμανικού Κοινοβουλίου. Το ρωτήσαμε τι έγινε. Αν υπήρξε πίεση. Όχι λέει πίεση. Μας έκανε συγκεκριμένες προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν μας έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Πράγματα που μας είπαν σε μισή ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας τα έχει δώσει σε 10 χρόνια. Αν θέλουμε λοιπόν μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, στην περίπτωση της Τιμοσέγκο, σε μια κρίση τέτοια, γιατί διαπραγματευόμαστε λοιπόν στην Ένωση αυτή, όταν τελικά είμαστε τόσο αποτυχημένοι και δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τον επόμενο προϋπολογισμό και η Ρωσία έχει 15 δισεκατομμύρια και τα προσφέρει μέσα σε μία ώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει στην πολιτική αυτή. Θα πρέπει λοιπόν σε μια νέα βάση να θέσουμε τη σχέση με την Ρωσία, να είμαστε, να συζητάμε με τη Ρωσία, να μην είναι αντίπαλοι μας. Ε, Mr. Stadler, Κύριε Στάντλερ, δέχεστε μπλε κάρτα. Παρακαλώ. Συνάδελφε Στάντλερ, ε, γνωρίζω τις τοποθετήσεις του κόμματός σας, της ομάδας σας και δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μου κάνετε εντύπωση γιατί τα ε, χρήματα του Ευρωπαϊκού Φορολογιουμενού θέλετε να, προσ... να διοχετευτούν προς Ανατολάς χωρίς όρους και σε τη φορά την ενδεχόμενη ε, προσχώρηση της Ουκρανίας. Αυτό έχετε υπόψη, δεν το έχω ακούσει κάτι σχετικό. Ε, Αδελφοί Λάμπστορφ, και εσείς ο ίδιος παραθέτω μίλησατε για παταγώδη αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της Ρωσίας. Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας, αλλά αν ξέρω εξ αρχής ότι κανείς δεν θέλει να χρηματοδοτήσει αυτή την ε, κατάσταση, γιατί προκαλώ τέτοια σύγκριση και ε, ε, αντίθεση, γιατί να αναμειχθώ στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Γιατί να προκαλέσω τέτοια σύγχυση αφού δεν ξέρω από την αρχή ότι δεν μπορώ να το πληρώσω αυτό. Δεν θα κάνω λοιπόν τέτοιο αγώνα κατά της Ρωσίας. Πιο σωστό είναι να κοιτάξουμε τι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και μετά να βρούμε έναν εταίρο στο διάλογο στο πρόσωπο της Ρωσίας και έχει έναν αντίπαλο. Κυρία ήταν ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, διάφοροι το ανέφεραν. Η Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία τρει ώρε διήρκησε την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό αποτυπώνει ουσιαστικά πόσο ψυχρό είναι το κλίμα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Ε, στο ψήφισμα το οποίο διαπραγματευθήκαμε χθε. Νομίζω ότι κάναμε αρκετέ συστάσει οι οποίε δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη βελτίωση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε ό,τι αφορά μια ενιαία φωνή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τη Ρωσία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι σχέσει είναι δύσκολε και ιδιαίτερα εν ώψη των γεγονότων στην Ουκρανία σε ό,τι αφορά την ασυμφωνία για τι εμπορικέ περιορισμού, τα θέματα για τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά το Σότσι και το καθεξής δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και διαπιστώνουμε ότι μετά από έξι χρόνια διαπραγματεύσεων ακόμα δεν έχουμε μια νέα συμφωνία εταιρική σχέση. Η σύνοδο δεν ήταν ελπιδοφόρο. Εκ παραλίλου θα ήθελα να πω ότι η Ρωσία ως γείτονα είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους μας και θα πρέπει να είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για όλη την περιφέρεια για όλη την πολιτική γειτονία, για την πρόεδρε. Αυτό που είναι καλό και για αυτούς, αλλά και για μας και για τους γειτονές μας. Και για να τα πετύχουμε αυτά θα πρέπει να συμβούν πιο πολλά, να γίνουν μεγαλύτερε προσπάθειες. Αυτά που λέει ο κ. Στάτλαν είναι λίγο απλοϊκά, θέλω να πω και να ρωτήσω, αυτά μπορείτε εσείς να τα πείτε και να τα πουλήσετε ε, στο εκλογικό σας κοινό. Όχι, ένα ανοιχτό διάλογο χρειαζόμαστε να θέσουμε τα προβλήματα επιτάπητος και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βρούμε κοινέ λύσεις σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Fleckstein, 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, η στρατηγική η εταιρική σχέση ορίζεται από κοινού στόχους και από κοινέ ευθύνε. Και σε, στις τρεις ώρες αυτές, στη Σύνοδο, προέκυψε το εξής. Πόσο απαραίτητο είναι και οι δύο οι πλευρές να συζητήσουν για τους στόχους αυτούς. Να αναζητήσουν τους στόχους αυτούς σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλέον, αλλά να συζητήσουν και για θέματα κοινής ευθύνης. Αυτό θεωρώ ότι δεν τονίστηκε αρκετά. Αλλά από την άλλη προέκυψε ότι μέσω της ε, κοινή συνθήκης ιστορικής σχέσης θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολλά πράγματα με καλή θέληση για πολλά θέματα της, κοινής, της πολιτικής ε, γειτονίας μπορούμε να διευκρινίσουμε τι ισχύει πραγματικά όπου υπάρχουν ανάγκες, όπου υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα και ένα κοινό project, ένα κοινό έργο, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δυστυχώς δεν μιλήσαμε για θέματα απελευθέρωσης θεωρήσεων. Αυτό δεν, είναι, δεν επιδεικνύει μεγάλη γενεοδορία. Και οι δύο πλευρές κάτι θέλουν να πετύχουν. Μεθαύριο ξεκινάνε οι αγώνες στο Σότσι. Χαίρομαι γιατί εκεί θα συναντηθούν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι και ελπίζω να περάσουν καλά όλοι μαζί. Και όταν θα ταξιδέψουν εκεί λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να τους πούμε είναι να μιλήσουν με τους νέους στη Ρωσία, να τους πούν τι γίνεται σε εμά. Να μιλήσουν με και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Να κάνουν ναι, ε, ομοφιλόφιλοι. Ό,τι και να είναι να μιλήσουν και νομίζω ότι αυτό θα το πετύχουμε, με αυτό θα πετύχουμε πιο πολλά από ότι με το ψήφισμα αύριο. Σας ευχαριστώ κύριο Λάμπστορ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, η κυβέρνηση στη ρωσικά λέγεται πρατσοβιτσικά, αλλά επίσημα κανείς ε, δεν ε, δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Γιατί η λέξη κυβέρνηση χρησιμοποιούν τη λέξη εξουσία. Αυτό καταδεικνύει και αυτό φαίνεται, αυτό δείχνει και το διακύβευμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Το θέμα είναι η εξουσία. Λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε τις ρητορικές. Να μην μιλάμε για μια στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι αντίπαλος, ανταγωνιστής ότι υπάρχουν θέματα στα οποία συνεργαζόμαστε, εντάξει, ναι, και για την ενέργεια και για την τρομοκρατία, αλλά πού είναι οι κοινέ αξίε, πού είναι οι κοινοί στόχοι που χρειάζονται για μια στρατηγική εταιρική σχέση, δεν υπάρχουν. Και η Ουκρανία είναι ένα κατεξοχήν παράδειγμα. Θα πρέπει λοιπόν νυφάλια να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Νυφάλια να μιλάμε με τις Ρώσους, να διαμορφώσουμε το status quo. Δεν μπορούμε να δώσουμε, να προσφέρουμε ε, προσχώρηση στην ε, Ουκρανία. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα status quo επωφελές για όλους. Χρειαζόμαστε εταιρική σχέση στην πολιτική, την εξωτερική. Χρειαζόμαστε προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικονομική συνεργασία. Οι στόχοι αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή μπορεί να συγκαταλέγονται στο πλαίσιο μιας εταιρική σχέσης. Σήμερα όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και η Ρωσία είναι μια ε, εξουσία που και για όλες τις συγκρούσεις ε, την Αυγαζία, την υπερπνευστερία, θέλει να τις αφήσει ανοιχτές. Δεν μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει μια τέτοια εταιρική σχέση. Θα πρέπει να είμαστε νυφάλοι και να διεξάγουμε διάλογο για να επιληθούν ένα-ένα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πιοτρόφσκι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Στο σχέδιο ψηφίσματος ε, της δικής μου ομάδα για την ε, Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, το πρώτο σημείο λέμε πως περιορίστηκε ε, η συμμετοχή σε αυτή την ε, ε, σύνοδο και μάλιστα περιορίστηκε και ο χρόνος στους οποίους, ο οποίος διατέθηκε στους συμμετέχοντες. Άρα λοιπόν δεν είχαμε πολύ χρόνο και δεν επιτράπη στους Ουκρανούς να έρθουν στην Σύνοδο. Και αμέσως μετά τη Σύνοδο είπαν οι Ρώσοι πως δεν θα δέχονται πλέον εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας τα λέω αυτά γιατί Θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο και την κυρία Άστον τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε ακολουθήσει μια παθητική στάση και ορίστε, ειδού τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Χόκμαρκ. Ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο. Um, Κύριε Πρόεδρε, η Ρωσία πρέπει να ανοίξει τα αρχεία της. Ε, ε, συμπεριλαμβανομένου του Ραλφ Βάλεμπεργκ. Γιατί ανοίγει ένα σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας έτσι. Δεύτερον, η Ρωσία θα πρέπει να παίξει πλήρως το ρόλο της ε, σαν εταίρος, αλλά δεν ενεργεί ως τέτοιος και αντίθετα απειλεί τους γειτονέ μας. Αυτό σημαίνει πως περιορίζει τις ίδιες τις ευκαιρίες να δράσει στην Ευρώπη, αλλά και να ωφεληθεί από την ε, εξάρτηση που έχουμε. Γιατί η εξάρτηση δεν πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτι αρνητικό, είναι μια ευκαιρία. Έχουμε εμπόριο, έχουμε μια ελεύθερη κυκλοφορία γνώσεων, διαχείρισης και όλα αυτά αυτά τα πράγματα που ε, περιλαμβάνονται στη συνεργασία. Τώρα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάπου, πρέπει να είμαστε πολύ ε, αυστηροί και σταθεροί για το γεγονός ότι η Ρωσία πρέπει να δεχθεί την κυριαρχία των γειτόνων της, να δεχτεί τα δικαιώματα των πολιτών της, να ζουν στη δημοκρατία και να δεχτεί ότι για να είναι εταίρος πρέπει να ενεργεί ως εταίρος μας. Ε, Δέχεστε μια μπλε κάρτα. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο Χόικμαρκ. Ο χάρτης ενεργειακός ε, για τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ κατέδειξαν ε, ότι υπάρχει καλή σχέση και για τις, δύο πλευρές που θα είναι αμοιβαία επωφελέ. Τι πιστεύετε για τις ενεργειακές ε, διαφορές μεταξύ τιμών, μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης. Αυτό στο μέλλον μπορεί να διαμορφώσει μια αποτελεσματική επιτυχή ιατρική σχέση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Εγώ πιστεύω πως η Ρωσία πρέπει να δεχτεί όλους τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά επίσης να, έχει, να είναι πιο λύση σε σχέση με την ενεργειακή της πολιτική. Από τη στιγμή που τη χρησιμοποιεί αυτή την ενεργειακή πολιτική ως έναν τρόπο για να επηρεάζει άλλες χώρες και άλλα έθνη και να ε, υπονομεύει τη δημοκρατία στα έθνη αυτά, Όσο το κάνει αυτό δεν θα έχει ποτέ τα πλήρη ωφέλη των πόρων της, των ίδιων αλλά ούτε και τη ωφέλη ε, των πόρων που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Θα πρέπει η Ρωσία να σεβαστεί βασικούς κανόνες σε σχέση με την οικονομία και να σταματήσει να επιβάλλει κυρώσει σε άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω περισσότερο για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Ρωσία. Έχουμε αυτές τις επιθέσεις από τον πρόεδρο Πούτιν που δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Επίσης, εναντίον των ομοφιλοφίλων, απαράδεκτο και ελπίζω πως οι αθλητές μας θα μιλήσουν στο Σότσι. Και βέβαια κατηγορώ και καταδικάζω τους χορηγούς όπως τη Βίζα, την Κοκακόλα, που ε, στηρίζουν αυτούς τους αγώνες. Εγώ θα τους μποϊκοτάρω και ξεκινώ με την Βίζα. Κυρία Πρόεδρε, όχι εξ ονόματός μου. Ευχαριστώ. Ε, Mr. Cashman, there is a blue card. Κύριε Κάσμαν, έχετε μπλε κάρτα. Ευχαριστώ πολύ που δέχτηκατε την ερώτηση. Εγώ στηρίζω το πολιτικό μποϊκοτάζ στο Σότσι, αλλά εκπλήσωμαι από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησατε σήμερα το πρωί, όταν η πολιτική μας ομάδα επέκρινε έναν από τους προέδρους για τον οποίο κάνει τις δουλειές τους, μας είπατε πως ε, την ε, επικρίνουμε για την γυναίκα και σήμερα μιλάτε για την ομάδα των ομοφιλοφίλων και τα λοιπά ε, που ε, υποτίθεται πλήττονται. Με συγχωρείτε, μπορούμε να το δούμε με κάποιο άλλο τρόπο και όχι ανάλογα με το γένος το θέμα. Εκτός μικροφώνου. Uh, Δέχομαι την ερώτηση του αξιότιμου μέλους, αλλά νομίζω ότι ήταν δήλωση. Δηλαδή, το να μην μιλάω για το φίλο πια ή για τις φυλετικέ διακρίσεις. Δεν θα πάψω ποτέ να μιλάω για τις διακρίσεις, οι οποίες έχουν ε, επιβληθεί σε κάποιους από αυτούς που θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα. Δηλαδή την τυραννία της πλειοψηφίας που προσπαθεί να καταπιέσει μια μειοψηφία. Να υπενθυμίσω ότι εσείς ζήσατε υπό την Σοβιετική κυριαρχία και την καταπίεση. Και οι αστικές ε, και οι κοινωνικές ελευθερίες και ο σεβασμός αυτών είναι το κατά είναι αυτό που αποφασίζει κατά πόσο κανεί είναι μια πραγματική και λειτουργική δημοκρατία. Εγώ λοιπόν δεν θα πάψω να μιλώ για αυτά τα ζητήματα. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Βοσιχόφσκι, ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις σχέσεις Ένωσης Ρωσίας δεν μπορούμε να ξεχνάμε τι συνέβη στις 10 Απριλίου 2011 στο Σμόλενσκ όπου συνετρίβει το αεροσκάφος με τον πρόεδρο Κατίνσκι που έχασε τη ζωή του της Πολωνίας και άλλους σημαντικούς αξιωματούχους. Ο λόγος για αυτή την καταστροφή δεν έχει ακόμα ε, εντοπιστεί. Συνεχίζονται οι έρευνες. Παρά τα αιτήματα της Πολωνίας, οι ρωσικές αρχές αρνούνται να φέρουν στην Πολωνία, να επιστρέψουν μάλλον στην Πολωνία το μαύρο κουτί που περιέχει έχει τα αρχεία του αεροσκάφους και αυτό θα ήταν απαραίτητο για να εξηγηθεί αυτή η καταστροφή. Γιατί το κρατάνε, γιατί αρνούνται να μας το δώσουν, αν και το έχουν στην κατοχή τους εδώ και τέσσερα χρόνια για να το αναλύσουν, για να το μελετήσουν. Εγώ πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαιτήσει αυτό το μαύρο κουτί καθώς και τα απομεινάρια του σκάφους για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το μυστήριο που κρύβεται πίσω από αυτήν την υπόθεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η κυρία Γιαννάκου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία δεν πάνε καλά. Αυτό είναι βέβαιο. Και δεν το δείχνει μόνο η τρίωρη συνάντηση, η οποία ήταν ελάχιστη. Ε, όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν για τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα, αλλά και την πρόσφατη ιστορία και τη θεωρία που φαίνεται να ισχύει αν δεν είστε μαζί μου είστε εναντίον μου. αλλά ας κοιτάξουμε από την πλευρά της ευρώπης. νομίζω ότι περιμένουμε περισσότερα από τη δική μας πλευρά. είναι μακρύτερη η ιστορία της δημοκρατίας και πιο σίγουρος ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε εμείς. εκεί υπάρχουν φόβοι και στη ρωσία και τις άλλες χώρες. πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο αν θεωρούμε ότι είναι αποδεκτό οι ηνωμένε πολιτείε να συνεργάζονται ως γενικός εκπρόσωπος της δύσης με τη ρωσία ή μέσα στην ευρώπη μεγάλες χώρες όπως η γερμανία να κάνουν το ίδιο τότε για ποια πολιτική ευρωπαϊκής ένωσης μιλάμε. αν θέλουμε πολιτική ευρωπαϊκής ένωσης που θα μετρήσει στη ρωσία και θα τη λάβει υπόψη της πρέπει να είναι η πολιτική της ένωσης και όχι η πολιτική των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σταμπαϊδη, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει λοιπόν να τιμήσουμε πραγματικά και με ρεαλισμό τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Δάλος θα ξεκινούσε ένας νέος ψυχρός πόλεμος κατά της ε, Ρωσία. Συμφωνώ με την κριτική, αλλά το ε, μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να δημορφωθεί χωρίς τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να μιλάμε υπόψη τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Η ρεαλιστική, βιώσιμα και αμοιβαία επωφελής στρατηγική σχέση, την οποία την οποία επέκριναν ε, άδικα ο κύριος Μπροκ δεν έχει, δεν αφήνει άλλη εναλλακτική και στην Ουκρανία. Θα πρέπει οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Ρωσία να ε, συζητήσουν και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με τη Ρωσία. Γιατί μιλάμε για μια τεράστια χώρα ε, στα σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μίλιαν Μόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που έγινε αυτή η Συνοδο ευρωπαικη Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία. Παρόλε τι διαφορέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αγνοεί μια γειτονική χώρα που είναι τόσο σημαντική με την οποία έχει τέτοιε ενεργειακέ και οικονομικέ σχέσει και εμπορικέ σχέσει, γιατί κάτι τέτοιο θα αυξήσει τα προβλήματα. Για μα είναι μεγάλο και παγκόσμιο παίκτη η Ρωσία και συστήθηκε μια ομάδα εργασία για τις συμφωνίες σύνδεσης στα πλαίσια της ε, εταιρική σχέσης ε, γειτονίας ε, και αυτό αποτελεί αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Πρέπει βέβαια να δούμε τι γίνεται και με τις χώρες επιρροής ε, της Ρωσίας. Θα πρέπει να σέβεται τις, την εθνική του κυριαρχία. Δεν μπορούμε να έχουμε νέα διέρεση στην Ήπειρό μας. Και ελπίζω τους επόμενους μήνες να προχωρήσει η διμερής επιτερική σχέση διαφορετικά ε, η Σύνοδος το μόνο που θα έχει κάνει είναι να χρησιμεύσει στην αντιτρομοκρατική μας συνεργασία. Θα πρέπει η συνεργασία με τη χώρα αυτή να είναι η συνεργασία εταίρων σε έναν πολυπολικό κόσμο που βρίσκεται μεταξύ Ευρώπης και Ασίας η Ρωσία θα πρέπει να βρει τον τρόπο να συνεργαστεί και μαζί μας όπως συνεργάζεται και με τους πέραν του Ατλαντικού εταίρους της. Δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από αυτό το μέλλον και νομίζω ότι για να το πετύχουμε θα πρέπει όλοι να σταθούμε ενωμένοι. Σας ευχαριστώ κύριο Σάιρος και για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία βρέθηκαν σε μια πορεία σύγκρουσης. Όταν η Ρωσία αμφισβήτησε ξαφνικά το πρόγραμμα Ανατολικής γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό προστέθηκε σε ήδη πολλά ανοιχτά, εκκρεμή ε, διμερεί ζητήματα. Η Ρωσία δεν μπορεί να δράσει και να ενεργήσει αντίθετα με τις ε, αξίες της ευρωπαϊκής αξίας και εκ παραλίλου να εκμεταλλεύεται το καθεστώς στρατηγικής συνεργασία. Το θέμα λοιπόν είναι, πρόκειται για σταθερή συνεργασία. Δεν υπάρχουν κοινοί στόχοι, δεν υπάρχει κοινή αξία. Ήταν ένα διάλογο μεταξύ κοφών στη Σύνοδο. Ε, η ρωσική επονίδηση πίεση στην Ουκρανία για να μην ξεκινήσει μια συμφωνία εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τελευταίο μήνα κατέστησε σαφέ ότι είναι πολύ αρνητική η στάση της Ρωσίας σε ό,τι αφορά την ανατολική πολιτική γειτονία και σε ό,τι αφορά την ε, Ουκρανία. Θα πρέπει η Ρωσία να μην αναμειγνύεται στα εσωτερικά της επικυρίαρχης ε, Ουκρανίας και να μην ασκεί τέτοια πολιτική πίεση. Κατά παραβίαση της ε, τελικής πράξης του Ελσίνκη και του memorandum του υπομνήματος του, για την απομάκρυνση των πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία. Προς μια τέτοια λύση λοιπόν θα πρέπει να οδεύσουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, ακόμα και οι αγώνες του Σότσκι δεν θα χαρακτηρίζονται από το πνεύμα που θα πρέπει να χαρακτηρίζονται της ε, συνεργασίας και της συμφιλίωσης. Grazie, onorevole Nitras. Un minuto. Ευχαριστώ, κύριος Νίτρας. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε μια θετική αξιολόγηση της πιο πρόσφατης αυτής συνόδου. Δεν μπορώ κι εγώ να συνταχθώ με τις απόψεις του Πρόεδρου Μπαρόσου, ο οποίος μας δήλωσε πως οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας αναπτύσσονται δυναμικά. Πρέπει να σου πω ότι ήταν μάλλον αφηρημένα τα όσα συζητήθηκαν στη Σύνοδο και δεν μπήκαμε σε απτά θέματα, για παράδειγμα τον αγωγό φυσικού αερίου, τα θέματα του ΠΟΕ, πρόσβαση στον αγωγό. Πρέπει να σας πω πως πολύ πρόσφατα είχαμε και ένα εμπάργο στην εισαγωγή χοιρινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας υπενθυμίσω πως πριν από 6 μήνες η Ρωσία απαγόρευσε τις εισαγωγές των ζωντανών ε, ζώων και των γαλακτονομικών στη χώρα. Μιλάμε για εμπορικό πόλεμο, όχι για φιλικές σχέσεις. Έχουμε κάποια εργαλεία για να την επηρεάσουμε, αλλά δεν έχουμε την τόλμη να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Και δεν είναι συμπτωματικό τότε ακόμα και τις δηλώσεις του Πούτιν τις δεχτήκαμε χωρίς κουβέντα ότι δεν θα μπορέσει ε, να δεχτεί ε, εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία η, Ρωσία γιατί οι ίδιοι δεν στέλνουν υπουργού να διαδηλώσουν στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Τι θα γίνει λοιπόν. Θα ακολουθήσουμε αυτή την τακτική και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νέινσκι, ένα λεπτό. Αξιότιμη κύριε και κύριοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, η σύνοδος αυτή έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η σχέση μας, τα συμφέροντά μας είναι υπερβολικά σημαντικά για να τα αφήσουμε στην άκρη και να μιλήσουμε τις διαφορές μας. Και οι διαφορές μας έχουν να κάνουν με την ανάγκη του να δεχτούμε την αρχή των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας θα πρέπει να απορρίψει αυτήν την ε, νοτροπία που επιβάλλει ε, από κοινού επιλογές χωρίς την δυνατότητα ο καθένας να ελιχθεί όπως χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα της Ουκρανίας και επίσης μια ενεργειακή πολιτική ευρωπαϊκή η οποία θα επιτρέψει στη Ρωσία να δεχτεί κάποιες πιέσεις μέσω αυτών των ενεργειακών μας σχεδίων. Η κοινή ενεργειακή πολιτική είναι σημαντικό εργαλείο και θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει ε, τα ε, εθνικά μας συμφέροντα. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποτινάξουμε και κάποια ιστορικά παραδείγματα. Bene, ci sono numerose richieste. Μάλιστα, πολλά αιτήματα κάτι έχω λάβει. Οπότε παρακαλώ να περιορίζεστε στο ένα λεπτό. Ο κύριος Στήρ. Κύριε Πρόεδρε, οι σχέσεις με τη Ρωσία ανέκαθεν ήταν και θα παραμείνουν κρίσιμες για την ασφάλεια της Ευρώπης. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη, ο πρώτος εμπορικός εταίρος ε, και η Ρωσία είναι ο τρίτος μας εμπορικός εταίρος, αλλά και άλλοι τομείς, όπως η καταπολέμηση του ε, της τρομοκρατίας, ε, η νοτιοανατολική Ευρώπη που για πρώτη φορά οι ρωσικές δυνάμεις μαζί με τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις με το ΝΑΤΟ ε, μπόρεσαν και ενήργησαν από κοινού το αποδεικνύουν. Ωστόσο η στάση της Μόσχας στην περίπτωση της Ουκρανίας αποδεικνύει πως η Ρωσία είναι έτοιμη να ενισχύσει τη θέση της, να την ενδυναμώσει εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων και κυρίως εις βάρος της κυριαρχίας ενός κράτους όπως η Ουκρανία και το δικαιώματο, εις βάρος του δικαιώματός του να αποφασίσει τι ρόλο και ποια πλευρά θα διαλέξει. Δεν θα πρέπει να διχαστούμε όμως ε, σε σχέση με την ε, Μόσχα, απέναντι μάλλον στη Μόσχα. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ κύριο Σκέλα μου. Όλες. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να, επινδε... να σας επιθυμίσω κάτι, ότι όσο τα κράτη-μέλη δεν ε, έχουν μια κοινή προσέγγιση, δεν θα έχουμε επιτυχή πολιτική για τη Ρωσία. Οι εξέλιξεις στην Ουκρανία μας εξαναγκάζουν να αναγνωρίσουμε ότι το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίπαλο, ε, ανταγωνιστή. Στην ε, ανομία που επικρατεί. Γι' αυτό λοιπόν ο στρατηγικό στόχο της Ρωσίας είναι να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση απαρνόμενη της ε, βάσης των αξιών της και δεν είναι πλέον κοινή η βάση των αξιών για να επιληθεί η κρίση με την Ουκρανία με επικοδομητικό τρόπο. Ο πρώτος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι να υπάρχει αρεσιμότητα. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε με την αναφορά και την διαβίβαση ισχυρών μηνυμάτων. Θα πρέπει καταρχάς ε, για παράδειγμα να παγώσουμε θεωρήσεις ε, για άτομα τα οποία ευθύνονται για διαφθορά και θα πρέπει λοιπόν αυτή να είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Κούκαν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αύριο ξεκινούν οι Ολυμπιακοί στο Σότσι. Είναι μια κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε σήμερα για τις διμερείς σχέσεις και για την κατάσταση ε, στη Ρωσία. Η σχέση μας με τη Ρωσία δεν είναι στη καλύτερη φάση της αυτή τη στιγμή. Αντικατοπτρίζει την συμπεριφορά της Ρωσίας εντός της ίδιας της επικράτειάς της αλλά και στις γειτονικές χώρες ε, η πίεση που ασκείται από τη Μόσχα στους γείτονές της είναι κάτι το παράδεκτο και μας θυμίζει τον νεοαπικιακό καθεστώς όπως ήδη αναφέρθηκε. Εξάλλου τα συμπεράσματα τη διάσκεψης κορυφή τη περασμένη εβδομάδα δεν μα εκπλήσουν. Είμαστε στρατηγική εταιρεία, αλλά έχουμε διαφορετικέ απόψεις και γνώμε για διάφορα θέματα όπω τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η Ουκρανία. Πρόθεσή μα και ανταπόκρισή μα στα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία δεν θα πρέπει να καθοδηγούνται από του Ολυμπιακού στο Σότσι. Όχι, είναι όμω μια κατάλληλη στιγμή ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί και διαυγής και να μιλήσουμε για τα όσα συμβαίνουν εκεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβούλιο, είναι η κατάλληλη στιγμή να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε, αλλά να βρεθούμε και σε μια κατάσταση όπου όλοι θα βγουν κερδισμένοι και είναι απαραίτητο αυτό να γίνει σήμερα με τη Ρωσία οι κυρώσει σε διεθνές επίπεδο δεν επιφέρουν αποτελέσματα γιατί αυτά σε πλήττουν τους πιο αδύναμους και τους φτωχότερους. Αντίθετα, οι αθλητικές ε, εκδηλώσεις αλλά και οι καλές οικονομικές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οι σχέσεις της Ρωσίας με το Ιράν είναι επίσης πολύ σημαντικές για μας. Ε, όμως οι κυρώσεις ενισχύουν τελικά ένα καθεστώς το οποίο στόχο έχει την αντιπαράθεση. Και εμείς οι Ευρωπαίοι οφείλουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα και όχι να επιβάλλουμε κυρώσεις, αλλά να θέσουμε τη συζήτηση στο επίκεντρο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Νεβεντάλοβα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανεί σήμερα ω προ το ότι χρειάζεται μια εταιρική σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία όμω θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν αμφισβητώ το γεγονό ότι η Ρωσία δεν εμένει πάντοτε στου όρου που από κοινού καθορίσαμε. Όμω και δικό μας φάλμα είναι, διότι ίσως και εμείς αλαζονικά σκεπτόμαστε. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να συνεργαστούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πήγα στη Μόσχα μία ημέρα μετά ε, την ε, διάσκεψη κορυφής ε, και σίγουρα όλοι ξέρουμε, έχουμε τις απόψεις για το τι συνέβη, γιατί ο τόσο γρήγορα, αλλά αυτή η πρώιμη λήξη της διάσκεψης κορυφής νομίζω έγινε αποδεκτή με ένα χαμόγελο από τη Ρωσία έρχεται μετά τον ψυχρό πόλεμο, εποχή των παγετώνων ε, στις σχέσεις μας, οι οποίες ε, γίνονται όλο και πιο ψυχρές και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό σε ό,τι δεν αφορά τους Ολυμπιακούς χειμερινούς αγώνες στο Σότσι. Πρόκειται για αθλητισμό. Δεν έχει να κάνει με την πολιτική αυτό το αθλητικό γεγονός και ο κόσμος ε, που έχει πάει εκεί θυσίασε χρόνια από τη ζωή του οι αθλητές. Ε, το να μην πάνε λοιπόν για πολιτικούς λόγους δεν έχει νόημα, διότι έχουν ε, προπονηθεί σκληρά για να εκπροσωπήσουν και τις χώρες τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρόμπεργκ. Η κυρία Η Ευρώπη έχει στρατηγικό εταίρο τη Ρωσία οι σχέσεις σε κρατικό επίπεδο δεν ε, δουλεύουν. Αλλά ενώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πρόβλημα με την κοινωνία των πολιτών. Ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα με την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία, θα πρέπει να δουλέψουμε και με τους νέους και με τους ακτιβιστές, να ενεργοποιήσουμε ανταλλαγέ ε, φοιτητών, νέων, ούτως ώστε να οικοδομήσουμε στο μέλλον αυτή την εταιρική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα μέσα για να το καταφέρει. Ευχαριστώ. Στίβενσον. Thank you very much, Madam President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ε, στη τηλεοράσεις σήμερα το πρωί εμφανίστηκε να προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ζωόφιλο κατά κάποιο τρόπο και καλό άνθρωπο ενώ ε, αδέσποτα ε, δολοφονούνται κατά εκατοντάδες στους δρόμους του Σότσι αυτές τις ημέρες. Δεν προεδρεύει όμως, αν θέλετε, μόνο στον τομέα της κατάχρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και κατά της κακοποίηση των ζώων. Είναι μάλλον ε, πρωταγωνιστής και στην κακοποίηση των ζώων. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εμεί, ξέρετε, σε συνδική τη Λισαβόνα, τα δικαιώματα των ζώων τα θεωρούμε σημαντικά. Ευχαριστώ. Όσο εντυπωσιακέ και αν είναι οι τελετέ ή τα γεγονόνα, τα, η χειμερινή Ολυμπιακή στο Σότσι θα βασιστούν, έτσι θα τη σημαίνει η ιστορία, θα βασιστούν στην ξενοφοβία, την εκμετάλλευση, τα σχόλια του Πούτιν για τους ΛΟΑΔ είναι προβληματικά. Ε, λέει ότι οκ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, φτάνει να αφήνουν τα παιδιά ήσυχα. Ένα περιβάλλον όπου η ομοφιλοφιλία θεωρείται έγκλημα και οι ΛΟΑΔ δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Έχουμε βία η εκμετάλλευση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, από εργοδότες που δεν πληρώνουν ε, τους μισθούς τους, τους κατάσχουν ε, τα διαβατήριά τους και τους αναγκάζουν να δουλεύουν 12 ώρες την ημέρα με μία μόνο μέρα ρεπό. Έτσι οικοδομούνται οι υποδομές του Σότσι. Θα θυμάστε τους Ολυμπιακούς του 1968. Είναι σημαντικό οποιαδήποτε πράξη προκλητική κατά των τάσεων αυτών στη Ρωσία να καλό είναι να της δοθεί ε, δημοσιότητα. Ο κύριος Σεβερίν. Η ευρωπαϊκή πολιτική προς τη Ρωσία είναι σχιζοφρενική. Αγνοούμε εντελώ το στρατηγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν οι σχέσεις μας. Και δεν αναγνωρίζουμε συγκεκριμένη ε, παράδοση, στρατηγική παράδοση της ε, Ρωσίας. Οι σχέσεις μας ε, επιδεινώνονται συνέχεια με τη Ρωσία γιατί επικρίνουμε συνέχεια την ε, γεωπολιτική της ε, στάση. Μην ξεχνάμε τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουμε ε, και δεν θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τη Ρωσία την τύχη των τρίτων χωρών ή να προωθήσουμε μαζικές πολιτικές. Εμείς μαζί με τη Ρωσία θα πρέπει να εναρμονίσουμε τις πολιτικές μας, να δείξουμε ενδιαφέρον για τις πολιτικές του του άλλου και για σεβασμό για τα δικαιώματα των γειτόνων μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τα στατηγικά μας συμφέροντα, συμφέροντα, αλλά να αναγνωρίζουμε και την πραγματικότητα. Δεν πρόκειται ποτέ η ευρωπαϊκή προοπτική από μόνη της να πριτανεύσει, εάν προωθήσουμε υπεριαλιστικές πολιτικές. Ας μην μιλάμε μόνο, ας μην έχουμε μόνο λόγια. Ας ε, στηρίξουμε τα λόγια μας με πολιτικές. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε το σεβασμό της Ρωσίας. Τελειώσαμε το Catch τώρα έχει το λόγο η Επιτροπή. Ο Επίτροπος Φιούλε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σκεφτόμουν πώς θα φαινόταν αν προσπαθούσα έτσι κάπως επιχειρησιακά ή τέλος πάντων να, στην πράξη να τα παρουσιάσω αυτά που άκουσα. Τρία σημαντικά σχόλια όμω θέλω να κάνω πρώτα απ' όλα σε σχέση με όσα είπαν οι Πρώτον, σε ό,τι αφορά αυτήν την ομάδα εργασία, οι ηγέτε συμφώνησαν στη διάρκεια τη ε, διάσκεψη κορυφή να δημιουργήσουν αυτή την ειδική ομάδα η οποία θα εξετάσει ε, τα αποτελέσματα που θα είχε η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ε, στα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα της Ρωσίας. Επιτρέψατε μου κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα, σε καμία περίπτωση δεν ε, παραβλέπουμε τους εταίρους μας στις συνομιλίες που έχουμε με τη Ρωσία, ούτε τους αγνοούμε. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Πρόκειται για συνομιλίες ε, γενικού περιεχομένου και δεν γίνεται λόγος για συγκεκριμένη εταιρική σχέση με συγκεκριμένη χώρα εταίρο. Δική μας πρόθεση είναι να συζητήσουμε τις ε, ρωσικές ανησυχίες που εκφράστηκαν. Σε δύο περιπτώσεις τη συνόψιζα. Πρώτον μετά τις ε, συμφωνίες ε, ελεύθερη DFCD, DCFTA, τα ευρωπαϊκά προϊόντα φοβούνται ότι θα κατακλείσουν τα, τις αγορές της χώρας εταίρου που έχει την Συμφωνία Ελεύθερου με την Ρωσία. Δεύτερο παράδειγμα, το οποίο αναφέρθηκε από τους Ρώσους εκπροσώπους, είναι ο ισχυρισμός ότι χρησιμοποιούμε την αγορά για τους εταίρους μας για επανεξαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων στις ρωσικές αγορές και στις αγορές της Ελληνιακής Ένωσης. Οι επιρρογνώμονές μας θα συζητήσουν ε, στη σχέση αυτή και στην ομάδα εργασία τα θέματα αυτά και θα τα εξηγήσουν ε, με απόλυτη σαφήνεια. Θέλω να σας πω ότι έχουμε ενημερώσει τους εταίρους μας για τη διάσκεψη αυτή και θα συνεχίσουμε να τους στηρούμε ενήμερους ε, για τις γενικές αυτές διαβουλεύσεις. Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές Εισαγωγέ και εξαγωγέ στη Ρωσία. Να καταστήσω σαφές και εδώ ότι αναλάβαμε δραστηριότητα, μιλήσαμε και ε, με, τους, ε, με τις υπεύθυνους στη Ρωσία, ο Μπόρκ, ο συνάδελφό μου, ο αρμόδιο για τα θέματα τη υγεία ε, και εγώ ανακοινώσαμε, κάναμε μια ανακοίνωση προηγούμενη Παρασκευή σε ό,τι αφορά τον πυρετό των χείρων. Αυτό δεν έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Η νόσος αυτή. Αλλά από τη Ρωσική Επικράτεια. Και πήγε και στη Λευκορωσία και μετά εξαπλώθηκε στην ε, Λιθουανία. Εμείς ε, λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίσουμε την εξάπλωση της νόσου σε ορισμένες περιοχές της Λιθουανίας με την λεγόμενη μέθοδο της περιφερειοποίησης και με τους ε, κανόνες ε, του ΠΟΕ και τα, τους ε, υγειονομικούς και φυτογειονομικούς κανόνες και πρότυπα που ισχύουν. και ελέγχουμε τις αγωγές εξαγωγές, ξέρουμε ότι έχουν ληφθεί δυσανάλογα μέτρα με τεράστιες επιπτώσεις για τη βιομηχανία μας. Το 25% των συνολικών μας εξαγωγών είναι εξαγωγές χειρίου κρέατος. Αν δεν βρεθεί λύση, θα ζητήσουμε να κινηθεί διαδικασία διαβούλευση σε επίπεδο ΠΟΕ. Αξιότιμοι βουλευτές, ε, θα δούμε, θα δούμε τι διδάγματα θα αντλήσει τώρα η Ρωσία και από τα γεγονότα της Ουκρανίας και από την ξεκάθαρη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή εκφράστηκε στη διάσκεψη κορυφής. Επιμένουμε ότι η συνεργασία θα πρέπει να εδράζεται στην αρχή του σεβασμού των κυρίαρχων αποφάσεων κάθε χώρα, των δημοκρατικών κοινωνιών, των ανοιχτών οικονομιών. Έχει συμφέρον, ισχυρό συμφέρον η Ρωσία να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται τι επενδύσει στην τεχνολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση παραμένει προσιλωμένη και στην υποστήριξη του εξυγχρονισμού τη Ρωσία. Ενδιαφερόμαστε πραγματικά για μια σύγχρονη, δημοκρατική, επιτυχημένη Ρωσία και εταιρική σχέση Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εξυγχρονισμό και η ανατολική εταιρική σχέση μπορούν να συμβάλλουν τα μάλα στο μέτωπο αυτό. Συζητήσαμε και το κοινό μας όραμα για ένα κοινό οικονομικό χώρο από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαντιβοστόκ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε ότι είναι πρόωρο να ξεκινήσουν τέτοιου είδου διαπραγματεύσει. Κατέστησε αυτή τη θέση τη. Αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι μια νέα συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Καλύτερη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις ε, τους στο πλαίσιο του ΠΟΕ και άλλες σημαντικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τήρηση των ε, σχέσεων που στην καλή γειτονία. Και τότε μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να αναπτύξουμε μια ισχυρότερη, βαθύτερη εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Θα πρέπει αυτή να είναι μια εταιρική σχέση που θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στο σεβασμό των ε, διεθνών δεσμεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Gracias, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτή με την παρέμβαση εκ μέρου ε, του Συμβουλίου του Προέδρου Βενιζέλου. Παρακαλώ κύριε Βενιζέλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις των αξιοτήμων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να τονίσω ότι σέβομαι και σεβόμαστε ως Προεδρία απολύτως όλες τις ευαισθησίες ευαισθησίες εθνικές ιστορικές γεωγραφικές αλλά και ευαισθησίες ιδεολογικές. ήταν πολύ επικοδομητική και επιβοηθητική η συζήτηση μετά την εμπειρία της πρόσφατης συνόδου κορυφής που σας την περιγράψαμε και ο επίτροπος ο κύριος Φίλε και εγώ. συμφωνούμε ως προεδρία με όλους εκείνους που θεωρούν ότι ως ευρωπαϊκή ένωση έχουμε μόνο μία επιλογή τη διαμόρφωση επικοδομητικών σχέσεων με τη ρωσία. η ρωσία δεν είναι ούτε εύκολος ούτε απλός εταίρος αλλά είναι αναγκαίος και κρίσιμος εταίρος. νέες διαχωριστικές γραμμές και νέες σφαίρες επιρροής στην ευρώπη πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθούν. θα ήμασταν απολύτως ανιστόρητοι εάν αφήναμε να εξελιχθούν τα πράγματα προς διληματικές ή διχαστικές καταστάσεις. αυτό θα ήταν αντίθετο τα συμφέροντα και της ευρώπης και της ρωσίας. η βελτίωση των σχέσεων ευρώπης ρωσίας θα αποβεί πολλαπλά επωφελής. δεν είναι μόνο το εμπόριο και οι επενδύσεις αυτές είναι σίγουρα θεμελιώδεις σχέσεις οι οποίες επηρεάζουν και τις πολιτικές μας κατευθύνσεις. συνεπώς τα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές πρέπει να καταργηθούν πρέπει να αυξηθεί ούτως ή άλλως αυξάνεται το διμερές εμπόριο υπάρχει μια θετική προοπτική υπάρχει προοπτική αμοιβαίων επενδύσεων πρέπει όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε εφόσον το μεγάλο μας πρόταγμα το μεγάλο ευρωπαϊκό πρόταγμα είναι η ανάπτυξη η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. υπάρχουν όμως και τα πολιτικά ζητήματα. δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη σύνοδο κορυφής και για την εταιρική σχέση ευρωπαϊκής ένωσης ρωσίας και να ξεχνάμε τα όσα έχουμε πει σε προηγούμενες συζητήσεις ακόμη και σήμερα στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για το πόσο κρίσιμη και αναγκαία είναι η συνεργασία ευρωπαϊκής ένωσης και ρωσίας για την εξέλιξη στη συρία για την εξέλιξη στο ιράν και την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος. είναι προφανές ότι όταν ασχολούμαστε με την εταιρική σχέση ευρωπαϊκής ένωσης ρωσίας συνυπολογίζουμε το πώς εξελίσσεται η σχέση ηνωμένων πολιτειών της αμερικής και ρωσίας όταν συζητούμε για τη σχέση ευρωπαϊκής ένωσης ρωσίας σίγουρα συνυπολογίζουμε το πώς εξελίσσεται η σχέση νατο ρωσίας και το συμβούλιο που λειτουργεί το συμβούλιο νατο ρωσίας. για να αξιοποιήσω μια παρατήρηση που έκανε η κυρία γιαννάκου προηγουμένως πράγματι πρέπει να δούμε ποια είναι η υπεραξία της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με τη ρωσία. προσωπικά μιλώντας έχω πολύ συχνά την εντύπωση ότι η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης σε σχέση με τη ρωσία είναι πολλές φορές μικρότερη από το άθροισμα των πολιτικών σχέσεων που έχουν τα επιμέρους κράτη μέλη διμερώς με τη ρωσία. χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή υπεραξία κάτι παραπάνω από το άθροισμα των διμερών σχέσεων με τη ρωσία και αυτό φαίνεται καθαρά σε πολλούς τομείς νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τομέας της ενέργειας. είχαμε την ευκαιρία στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων στην αφετ να συζητήσουμε πιο αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. έχουμε μπροστά μας ορισμένα εργαλεία που πρέπει να αξιοποιήσουμε πέρα από την εντατικοποίηση των εμπορικών συναλλαγών είναι η σύναψη μιας πιο φιλόδοξης ολοκληρωμένης νέας συμφωνίας. υπάρχει πάντα το ζήτημα της διευκόλυνσης των θεωρήσεων εισόδου κάτι που αφορά ιδιαίτερα τους τουριστικούς προορισμούς στην ευρώπη και τελικά την απελευθέρωση των θεωρήσεων μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. πρέπει να πετύχουμε πρόοδο στα θέματα αυτά έχοντας φυσικά πάντα υπόψη μας το στρατηγικό πλαίσιο των σχέσεών μας. πρέπει να αφιερώσουμε πολλές ώρες συζήτησης και στο συμβούλιο και στο κοινοβούλιο για το στρατηγικό πλαίσιο και τις ισορροπίες και πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή ήδη έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να καταγραφούν εξαιρετικά χρήσιμε απόψει που σημείωσα για να μεταφέρω στο συμβούλιο που θα συζητήσει πολύ σύντομα ξανά για τις σχέσεις ευρωπαϊκής ένωσης ρωσίας. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος για την ολοκλήρωση της ε, συζήτησης αυτής. Βέβαια τώρα λίγη συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο το μεσημέρι. Επί των προτάσεων αυτών ψηφίσματος. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο αφορά δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με οι καζόμενες αποθήσεις στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών